Bonjour à tous. Χαίρετε και καλώς ήλθατε στη συνέντευξη τύπου. Θα σας ε, παρουσιάσω την Άννη Ποδηματά, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου και εισηγήτρια για την έκθεση για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και κοντά της είναι η κυρία Γκρίφις Jones, γνωστή οικονομολόγος, η οποία με τον κύριο Άπενας Περσό συνυπογράφει μελέτη για την επίπτωση του φόρου, τι επιπτώσει μάλλον του φόρου των χρηματοπιστικών συναλλαγών και αντίγραφα θα βρείτε στο πίσω μέρος της αίθουσα Μετά από την συνέντευξη αυτή τύπου η κυρία Γκρίφης Τζόνς θα συμμετάσχει σε ακρόαση της Οικονομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Το λόγο θα λάβει αμέσως η κυρία Ποδηματά και αμέσως μετά η κυρία Γκρίφης Τζόνς θα πει λίγα λόγια δηλαδή για τα βασικότερα συμπεράσματα της ε, μελέτης της και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ Σολάνς, σας ευχαριστώ και όλους που ε, παρευρίσκεστε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ όλος ιδιαίτερος την κυρία καθηγήτρια Griffith Jones που βρίσκεται σήμερα μαζί μας και που μαζί με τον κύριο Άβινα Περσό, ο οποίος ε, λόγω χιονιού δεν μπόρεσε να προσέλθει, συνυπογράφουν την καλοθεμελιωμένη αυτή αξιόπιστη και περιεκτική μελέτη για την εφαρμοσιμότητα, το σωστό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όπως εξηγήσει η ειδικό μας, η μελέτη αναφέρεται σε συγκεκριμένες πτυχές της πρότασης της Κομισιόν για κοινό σύστημα εφόρων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, πρόταση η οποία όπως ξέρετε δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο Οκτώβρη σε ανταπόκριση πλειώνων εκκλήσεων του Κοινοβουλίου για παράδειγμα δύο ψηφίσματα του Μαρτίου 2010 και του Μαρτίου 2011 όλα ε, αυτά τα ψηφίσματα συνταγμένα από εισηγητές της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Για τις τεχνικές πτυχές της προτάσεως που θα επισέλθουμε περισσότερο και θα ε, διερευνήσουμε τις δυνατότητες βελτιώσεως. Εκτός λοιπόν από αυτές θεωρούμε ότι στο σύνολό της η πρόταση της Κομισιόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση διότι υποστηρίζει και υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τη λογική που εμείς έχουμε υποστηρίξει από πολύ καιρό για την εισαγωγή του φόρου αυτού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας παγκόσμιας συμφωνίας. Ο οποιοδήποτε σχετικός φόρος που θα πρέπει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογής, φόρος δηλαδή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και με χαμηλά, χαμηλούς συντελεστές θα εξασφαλίσει ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμβάλλουν για το ξεπέρασμα της κρίσης, να μειώσει τον κατακαιρματισμό, να ε, τονώσει την εναρμόνιση και τη συνεργασία στην ενιαία αγορά και με την ευκαιρία αυτή τονίζω ότι αν όντως θέλουμε μια ισχυρότερη, πιο ενοποιημένη και λιγότερο ε, διαστρεβλωμένη ενιαία αγορά, όπως άλλωστε πολλοί έχουν πει τους τελευταίους μήνες, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει κατ' επιλογή, με μια επιλεκτική προσέγγιση à la Νομίζω ότι θα έπρεπε και μπορούμε άλλωστε, εκτός και από άλλα κίνητρα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόσφατα εγκεκριμένο ρυθμιστικό καθεστώς και καθεστώς εποπτείας, με όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία μπορούμε να δώσουμε μπορούμε να μειώσουμε, να δώσουμε αντικίνητρα δηλαδή στην κατάχρηση ορισμένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών οι οποίες υποσκάπτουν εν τέλει την οικονομία και δεν τις προσφέρουν ρευστότητα. Όπως λέει η μελέτη και όπως θα εξηγήσει η κυρία καθηγήτρια σε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες, θέλουμε να κάνουμε αυτή την ανεπιθύμητη δραστηριότητα που περιέχει και υψηλό ρίσκο αλλά χαμηλή απόδοση να γίνει υψηλή απόδοσης και χαμηλού ρίσκου. Αυτό θα έχει άλλωστε ευεργετική επίδραση στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, θα ενθαρρύνει και δεν θα αποθαρρύνει όπως ε, ισχυρίζονται οι αντίπαλοι του φόρου και τις επενδύσει αλλά και την απασχόληση στην Ευρώπη. Και εν τέλει και ως συνέχεια των συμπερασμάτων της πιο, του πιο πρόσφατου άτυπου Συμβουλίου της 23 η Ιανουαρίου που έριξε ιδιαίτερο βάρος όπως γνωρίζετε στην οικονομική, στη δημοσιονομική μάλλον εξυγίανση που να είναι ωστόσο φιλική προς την ανάπτυξη και που περίλαβε ωστόσο ακόμα αυστηρότερα μέτρα για την δημοσιονομική εξυγίανση χωρίς να περιλάβει μέτρα για την πρόθεση της ανάπτυξης. Αντί για αυτά λοιπόν εμείς θα προτείνουμε μια προσέγγιση φιλική στον πολίτη μια προσέγγιση η οποία να θέσει τα θέματα της δημοσιονομικής εξυγίανσης χωρίς ωστόσο να, βάλει, να φορτώσει όλα τα βάρη στον απλό φορολογούμενο. Μια δηλαδή προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει και ειδικά μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης. Και εμείς πιστεύουμε ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας προσέγγισης. Ευχαριστώ πολύ και Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Στέφανη Γκρίφις Τζόουνς η οποία θα μπορέσει να μας εξηγήσει τα πιο σημαντικά στοιχεία της ε, μελέτης που έχει συνυπογράψει μαζί με τον κύριο Πέρσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία που μπορώ να λάβω το λόγο αμέσως μετά τη θαυμάσια εισαγωγή της Άννη Ποδηματά που ξεκαθάρισε το λόγο που δικαιολογεί ε, την επιβολή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και άλλωστε το κείμενο της Κομισιόν τονίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση της οικονομικής κρίσης και το λόγο αυτό θα πρέπει να συμβάλλει με δικαιότερο τρόπο στην επίλυση της κρίσης και στην ανάκαμψη. Και είναι σημαντικό επίσης να τονίσει κανείς ότι ο χρηματοψηφικό τομέα είναι πολύ λίγο φορολογημένο. Δεν πληρώνει, για παράδειγμα, ΦΠΑ. Ελάχιστοι τομεί οικονομία δεν το πράττουν. Επίση, για να ενθα... ενθαρρύνει αυτή η πρακτική, ενθαρρύνεται μάλλον αυτή η πρακτική, η οποία εμπεριέχει σημαντικό ε, ρίσκο. Και αυτό βέβαια θα είναι ένα συμπληρωματικό αποτέλεσμα, η αποθάρρυνση δηλαδή. Ήθελα να πω επίση με λίγα λόγια ότι συχνά ο ίδιο ο χρηματοπιστωτικό τομέα ισχυρίζεται ότι η ιδέα του φόρου αυτού είναι ε, κακομασιμένη. Ωστόσο ο ίδιος ο Κέινς που πολλοί οικονομολόγοι θεωρούμε ότι ήταν ο μεγαλύτερος οικονομολόγος, οικονομολόγος του προηγούμενου αιώνα αυτός στην αρχική του θεωρία τον προτείνει, τον έχουν υποστηρίξει και πολλοί νομπελίστες όπως ο Τόμπιν, ο Στίγλιτς με τον οποίο είχα την, τη χαρά να συνεργαστώ και άλλοι κορυφαίοι όπως ο Ήπλος, Ευρωπαίοι οικονομολόγοι έχουν υποστηρίξει το φόρο αυτό. Αυτά όμως, ε, δεν είναι όμως μόνο πανεπιστημιακοί αυτοί που τον έχουν υποστηρίξει αλλά και άνθρωποι της πράξης που έχουν ωστόσο κορυφαίο ρόλο στον ε, χρηματοοικονομικό κόσμο. Για παράδειγμα, ο Λόρδος Τέρνερ της Βρετανικής ε, Αρχής Εποπτείας που λέει καθαρά ότι θα είναι καλό πράγμα να επιβληθεί ο, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο δε συνυπογράφων που ε, έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στο City του Λονδίνου, επίσης υποστηρίζει την ιδέα αυτή. Γιατί τώρα ο φόρος αυτός είναι μια ιδέα που έχει έρθει πια η ώρα της σήμερα μέσα στον αγώνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει, η Ευρώπη μάλλον να ξεπεράσει την κρίση. Έχει πολλά οικονομικά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα αυξήσει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα. Πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μια εποχή που γνωρίζουμε όλοι ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγάλα ελλείμματα και χρέη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή μερικώ για ορισμένε χώρε για την εξυγένση των οικονομικών του. Αυτό είναι λίγαν επιθυμητό. θα μειώσει το κόστο δανεισμού των κυβερνήσεων και αυτό είναι πολύ θετικό για να εξασφαλίσει ανάπτυξη και θα μειώσει κάπως τη σοβαρότητα της κρίσης του χρέους. Με τη μείωση του ελλείμματος θα επιτρέψει να αυξηθούν και οι ιδιωτικές επενδύσεις και αυτό ασφαλώς είναι πάρα πολύ θετικό. Ένα άλλο, μια άλλη ενδεχόμενη χρήση του, ε, του φόρου αυτού που έχει ιδιαίτερη σημασία πάλι σήμερα μέσα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο της υψηλής ανεργίας των χαμηλών επενδύσεων και τη ανάγκη να γίνουν επενδύσει στην πράσινη οικονομία γιατί ο πλανήτη δεν μπορεί να περιμένει πλέον. Έτσι λοιπόν ο FTT εν συντομία στα αγγλικά μπορεί είτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ε, υλοποιηθεί αυτό είτε από τι χώρε μέλη μπορεί να χρηματοδοτήσει αύξηση των επενδύσεων για πράσινη υποδομή, για ανανεώσιμε ενέργειες ή για να παίξει ρόλο καταλήτη για επενδύσεις στις ε, καινοτομίες από πλευράς μικρών και μεσών επιχειρήσεων και να δημιουργήσει έτσι ανάπτυξη. Θα έχει λοιπόν και βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα που ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για την τόνωση της ζήτησης αλλά θα έχει και ε, ε, αποτέλεσμα και από την πλευρά της προσφοράς. Ορισμένοι από τους πόρους αυτούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εμέσως, δηλαδή μπορεί να αυξηθεί το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης και μπορεί να αυξήσει έτσι τον δανεισμό που προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα. Και επομένως ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η επίδραση, αφού έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα λόγω της μόχλευσης, στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι και ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεση ή χαμηλής ανάπτυξης, μπορεί αυτός να αποδειχθεί ιδεώδη τρόπος για την αύξηση τη ανάπτυξη, διότι ο ιδιώτης επενδυτή είναι πολύ ανήσυχο λόγω τη χαμηλή ζήτηση και ούτω καθεξής και της αβεβαιότητας. Αν λοιπόν διοχετευθούν τέτοια δημόσια ε, κονδύλια, αυτό θα βελτιώσει και μπορεί να οδηγήσει, τρίτο αποτέλεσμα, να μειωθούν άλλοι φόροι. Έχουμε σημαντικά πάντως στοιχεία και από πλευράς Κομισιόν και από αλλού ότι ο FTT θα είναι προοδευτικότερος από άλλους φόρους και μπορεί να σημάνει ότι ένα υψηλότερο ποσοστό του ε, μεριδίου εισοδημάτων των φτωχότερων νοικοκυριών θα καταναλώνεται διότι οι φτωχότεροι, ως γνωρίζετε, καταναλώνουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους από ότι αναλογικά οι πλουσιότεροι. Άρα οι investment managers θα έχουν λιγότερα λεφτά στη διάθεσή τους, αλλά οι νοικοκυρές περισσότερα. Άρα αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ε, ζήτησης και άρα της ανάπτυξης. Ορισμένα από τα επιχειρήματα κατά του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από τα πρώτα που προβάλλονται είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και ότι θα έπρεπε να αποφευθεί. Εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι στην πρώτη διάσκεψη όταν συζητήθηκε ο νόμος Τόμπιν. Και ο Τόμπιν είπε όταν προ εκατοντάδων ετών εισήχθη ο φόρο εισοδήματο, το πρώτο σχόλιο που έκανα είναι όλοι, άμα θα γίνει φοροδιαφυγή. Και βεβαίω έγινε φοροδιαφυγή. Αλλά εξακολουθεί να αποδίδει 500 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ, υποθέτω. Και επομένω μπορεί να επιβληθεί όπω κάθε ε, φόρο και θα αποδώσει. Δεύτερο, έχουμε καλά επιχειρήματα, έχουμε μάλλον ε, θαυμάσια παραδείγματα φόρων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που λειτουργούν, που αποδίδουν. Και ο καλύτερος είναι ο Βρετανικός stamp duty, φόρος χαρτοσύμου δηλαδή, που έχει αποδώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και εκεί η φοροδιαφυγή είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Να λοιπόν ένα θαυμάσιο παράδειγμα ενός επιτυχούς φόρου που βασίζεται τη στιγμή, μα που εισπράτεται μάλλον ή που γίνεται εισπρακτέως στη στιγμή που νομιμοποιείται η συναλλαγή. Και η συναλλαγή δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν εισπραχθεί ο φόρο. Άρα ο ουδής μείζων επενδυτής δεν θα αναλάβει τον κίνδυνο να μην καταβάλει ένα ελάχιστο φόρο ώστε να έχει κάποιο όφελος. Αν θέλει για παράδειγμα να επαναπολύσει τη συναλλαγή. Και αυτό βέβαια δεν είναι, δεν είναι μόνο η περίπτωση του Βρετανικού stamp duty, υπάρχουν και άλλοι, για παράδειγμα στην Ινδία, το Hong Kong, τη Σεούλ, που είναι και από τα κέντρα μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα επιχειρήματα εδώ. Και τέλος, θέλω να έρθω και στο πιο πρόσφατο επιχείρημα κατά του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που λέει ότι θα αποβεί κακός για την ανάπτυξη. Στο κείμενό μας έχουμε προβεί σε λεπτομερή ανάλυση βασισμένη σε ένα μοντέλο του ονόσων έχει ε, φτιάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούμε ότι ο FTT, καταλήγουμε στο ότι ο FTT μάλλον θα αυξήσει το ΑΕΠ. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο το κάνουμε αυτό είναι διότι ένα πολύ μικρό μέρος της χρηματοδότησης των επενδύσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως δείχνει και το πιο πρόσφατο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόνο λοιπόν ένα μικρό μέρος, 15% θα φορολογείται, διότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων χρηματοδοτείται είτε από επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια ή από επιστροφές φόρων. Ένα πολύ μικρό λοιπόν ποσοστό, μόνο 15% από αυτές θα βαρύνεται από τον ε, FTT. Και ένα μεγάλο μέρος του φόρου, όπως επιχειρηματολογείο Τόμπιν και άλλοι θα επιβάλλεται σε trading μεγάλης συχνότητας που δυστυχώς φτάνει τώρα το 40% των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αν λοιπόν αυτές οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας μειωθούν, αυτό θα αποδειχθεί καλό, διότι αυτές οι συναλλαγές έχουν αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, εάν υπάρξει ένα πρόβλημα ρευστότητας, αφαιρούν ρευστότητα οι συναλλαγές από το σύστημα, όπως έγινε το Μάιο του 2010 στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών των τροποποίησεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μελέτη της θεωρεί ότι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι τη τάξη του 0,1% του ΑΕΠ. Αλλά δεν λαμβάνει υπόψη ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του FTT ότι θα μειώσει δηλαδή τον κίνδυνο μελλοντικών κρίσεων. Και η εκτίμηση που κάνουμε είναι πολύ συντηρητική, διότι υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει η ε, νομοθεσία πρόληψης και άλλες μακροοικονομικές πολιτικές. Εμείς λέμε ότι η FTT θα μειώσει κατά 5% λένε μόνο τη ε, πιθανότητα μελλοντικών κρίσεων. Και έχουμε ένα πρόσθετο ε, αποτέλεσμα 3,5% του ΑΕΠ. Έχουμε λοιπόν ένα 0,25% του, ε, του ΑΕΠ ως πρόσθετο αποτέλεσμα. Και ο Τόπι λέει ότι αν μειωθούν λίγο τα σχετικά έσοδα των ε, όσων ασχολούνται τον χρηματοπιστωτικό τομέα θα προσελκύσετε και άλλους να ευφύς ανθρώπους νέους να πάνε και αλλού, δηλαδή στην έρευνα και ούτω καθεξής και να γίνει πιο παραγωγική η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί λιγότερο παραγωγική. Ε, real engineering, δηλαδή πραγματική μηχανική αντί για τους financial engineers. Και αυτό θα είναι βέβαια ευεργετικό για τη μελλοντική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Και το τελευταίο που λέμε είναι ότι ο FTT δεν θα οδηγήσει μόνο σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά σε καλύτερη ποιότητα ανάπτυξη θα βελτιώσει, δηλαδή θα κάνει την ανάπτυξη λίγο πιο δίκαιη και αυτό είναι καλό διότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβολική συγκέντρωση εισοδήματος και πλούτου και θα την κάνει πολύ πιο πράσινη και βιώσιμη και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Άρα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερη ανάπτυξη, δηλαδή πιο ισότιμη και πιο ε, βιώσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Ρεμπέκα Κρίστη από το Down News. Μήπως έχετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα φόρων τα οποία ε, μπορούν να περικοπούν ή να μειωθούν. Αν υπάρχουν προτάσεις για να γίνουν τέτοια ανταλλαγέ φόρων όπως περιγράφεται απάντηση, αυτό κοιτάξτε είναι πολιτική απάντηση, αλλά για παράδειγμα στη μείωση του ΦΠΑ που σε γενικά που γενικά είναι πιο επιθετικό. Το έχει προτείνει κανείς, το έχει προτείνει κανεί σε καμία χώρα, ερώτηση, απάντηση. Νομίζω ότι, ότι η γενική γραμμή είναι προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής ε, ενοποίησης για τη μείωση των ε, χρεών και των ελλημάτων, το οποίο στο πλαίσιο της κρίσης θα ήταν πολύ χρήσιμο. Florence je suis tout ici à droite, madame. Uh, uh, Εδώ είμαι. Στα αγγλικά δεν φοβάστε ότι θα δημιουργηθεί, θα δημιουργηθεί ένα δίλημα για τις κυβερνήσεις, γιατί εκ παραλλήλου υπάρχουν και οι συστημικοί κίνδυνοι και παράλληλα προσπαθούμε να ε, κερδίσουμε κάποια χρήματα για τους εθνικούς ε, προπολογισμού. Μήπως ε, υπάρχει τάση για πιο πολλές συναλλαγές, γιατί πιο πολλές συναλλαγές θα ευνοήσουν και τον φόρο των συναλλαγών και αυτό λένε κάποιοι εμπειρογνώμονες, ότι σκοπός του φόρου δεν είναι να μειωθούν οι συναλλαγές και ο συστημικός κίνδυνος, αλλά να συλλεχθούν χρήματα. Είναι σωστό αυτό. Υπάρχει τέτοιο δίλημα. Απάντηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο δίλημα, γιατί ο φόρος αυτός θα είναι χαμηλός και θα έχει υψηλή απόδοση ακριβώς επειδή υπάρχουν τόσες πολλές συναλλαγές θα υπάρχει κάποια μείωση των συναλλαγών, αλλά αν θέλετε στις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, το οποίο είναι και η αρχική φιλοσοφία. Για παράδειγμα, ένα τρέιντερ υψηλής συχνότητας θα πληρώνει εκατονταπλάσιο φόρο από ένα ταμείο συνταξιοδότησης, γιατί ένα ταμείο συνταξιοδότησης ε, αγοράζει μετοχές ε, μία φορά στα δύο χρόνια, ενώ ο trader, για παράδειγμα, κάθε μέρα, κάθε ώρα ίσως. Άρα, προφανώς ε, το γεγονός ότι θα, θα προκληθεί μία αποθάρρυνση σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές θα αφορά μόνο τους, ε, ε, αυτούς που κάνουν πολλές συναλλαγές και επίσης θα έχει υψηλή απόδοση, δηλαδή θα μαζεύονται πολλά χρήματα το οποίο θα επιτυγχάνει και τους δύο στόχους μας. Αν ε, είναι κανείς μακροπρόθεσμος ε, επενδυτής δεν θα επηρεαστεί αν για, κατα... για παράδειγμα κατασκευάζει κανείς ένα εργοστάσιο, δεν τον αφορά καθόλου. Στα γαλλικά. Ε, έριξα μια ματιά μόνο στην μελέτη σας. Αν κατάλαβα καλά, αναγνωρίζετε ότι η αρχή της διαμονής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα εμποδίσει να υπάρξουν μετακινήσεις εδρών καταστάσεις δηλαδή, δηλαδή επιχειρήσεων και αναφέρεστε και στο παράδειγμα PSA, μπορείτε, δηλαδή της Peugeot Citroën, μπορείτε να εξηγήσετε με περισσότερες λεπτομέρειες. Απάντηση. Αυτό που προτείνουμε είναι ένας συνδυασμός και των δύο προσεγγίσεων, ώστε να είναι πιο συνεκτική Δηλαδή αυτό το stamp duty, όπως ο φόρος χαρτοζήμου ο Βρετανικός, που επιβάλλεται και στους αλλοδαπούς. Πάρα από 40% του Βρετανικού stamp duty, stamp duty επιβαρύνει αλλοδαπούς. Αλλά συμπληρωματικά θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια αρχή που προτείνεται από το, από το σύστημα της Κομισιόν δηλαδή και τους ημεδαπούς αυτούς που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα για τις συναλλαγές τους στην αλλοδαπή. Αυτό θα είναι το σύστημα καλύτερο διότι θα είναι πιο συνολικό, πιο περιεκτικό. Προδηματά. Τονίζω ακόμη ότι αυτή είναι η προσέγγιση που σκοπεύει να ακολουθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ένας συνδυασμός της αρχής της residence όπως προτείνει η Κομισιόν αλλά και της issuance διότι αυτή είναι η πρώτη μας ε, εντύπωση, αυτή η πρώτη μας ε, σκέψη ότι αντιμετωπίζεται σωστά έτσι με το residence principle δηλαδή το θέμα των παραγόγων ενώ το άλλο δηλαδή του τόπου εκδόσης είναι για τα υπόλοιπα είναι ωστόσο μια δυνατότητα αυτή να μειωθεί και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε κάπως να βελτιώσουμε δηλαδή την άνηση μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις ευρωπαϊκές, στα ευρωπαϊκά αξιόγραφα που θα, ήταν, είναι καλύτερο επομένω από το εάν υιοθετηθεί όπως έχει η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται μόνο στην αρχή της, του τόπου διαμονής. Νομίζουμε λοιπόν ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών αρχών θα ε, βελτιώσει, θα εξασφαλίσει μάλλον καλύτερη εφαρμογή του φόρου και ταυτόχρονα θα είναι πολύ πιο δίκαιη αφού θα καλύπτει όλα τα είδη των συναλλαγών αλλά και φορέων που συναλλάσσονται στη βάση ε, ευρωπαϊκών assets, ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων. Για τον Ουγγρικό τύπο, θα ήταν καλή ιδέα να εισαχθεί αυτό ο φόρο επί των χρηματιστικών συναλλαγών σε μία μόνο χώρα, στη Γαλλία για παράδειγμα, ή σε περιορισμένο ρυθμό ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί βλέπουμε πώ εξελίσσονται οι συζητήσει και προ ποια κατεύθυνση κινούνται και δεν υπάρχουν πολλέ ελπίδε ότι θα εισαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απάντηση, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ερώτημα. Προφανώ, ε, ιδανικά, θα πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά. Αλλά αν έτσι δεν καταλήξουμε σε διεθνή συμφωνία και δεν περάσει ο φόρος, το να περάσει σε μία χώρα και να καταδείξουμε ότι δουλεύει και μάλιστα ε, έχουμε διάφορες χώρες που το έχουν εισάγει σε περισμένο βαθμό, όπως η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν εισαχθεί λοιπόν σε μια χώρα ε, όπως η Γαλλία, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό προηγούμενο για άλλες χώρες και θα καταλάβουν και οι άλλες χώρες, αν πάνε όλα καλά, ότι θα πρέπει και αυτές να τον εισάγουν. Φυσικά πολύ καλύτερο θα ήταν να εισαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η ευρωπαϊκή αγορά είναι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο. Αλλά αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι η εθνική εφαρμογή είναι ένα θετικό βήμα και είναι επίσης θετική η ιδέα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ο φόρος αυτός αν εισαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να περάσει από αξιολόγηση και εκτίμηση μετά από τρία χρόνια γιατί πάντα γίνονται συζητήσεις αλλά γιατί να μην το εφαρμόσουμε, να δούμε πώς λειτουργεί και μετά να δούμε πώ μπορούμε να το βελτιώσουμε. Έτσι γίνεται με τι οικονομικέ πολιτικέ. Η κυρία Ποδηματά. Ναι, συμφωνούμε ασφαλώ ότι η καλύτερη επιλογή για την εισαγωγή του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι σε καθολικό επίπεδο. Αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Επιμείναμε άλλωστε στην ιδέα εισαγωγής ενός τέτοιου φόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο επειδή πιστεύαμε ότι κάποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Αν πραγματικά θέλουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, όπως και να έχει σήμερα, έχουμε διάφορες επιλογές για το... Μάλλον υπάρχουν και εφαρμόζονται διάφορα είδη τέτοιου φόρου σε διάφορες χώρες. Δηλαδή, όπως αναφέρθηκε στον Εμμένο Βασίλη αυτό το τέλος χαρτοσύμου. Αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές τέτοιου φόρου επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που εφαρμόζονται ήδη. Θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματεύτηκε διάφορα τέτοια παραδείγματα φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που ήδη έχουν εφαρμοστεί σήμερα ή που έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν όπως ήταν ο περίφημος σουηδικός φόρος και νομίζω ότι έχουν βγάλει και κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τις διάφορες στρεβλώσεις που ε, δημιουργήθηκαν μετά από κάποιες μορφές τέτοιων φόρων, λαμβάνοντας υπόψη και το τι λοιπόν ε, έγινε με τους ε, διάφορους φόρους που ίσχυσαν ή ισχύουν σήμερα ακόμη. Άρα ανάλογα με τις εμπειρίες αυτές και τα πορίσματα αυτά προτάχθηκε η σημερινή αυτή πρόταση. Να υπενθυμίσω κάτι που είπα και εισαγωγικά, ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τον κατακριματισμό της ενιαίας αγοράς σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές αλλαγές που αποτελεί και ουσιαστικά την αιτία της κρίσης και νομίζω ότι αυτό είναι βασικό κρίσιμη σημασία αν θέλουμε να περιορίσουμε τους συστημικούς κινδύνους και επίσης είναι απόλυτα απαραίτητο αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και να την καταστήσουμε πιο ενοποιημένη. Αυτό ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπέρ μια, μιας πιο ισχυρής ε, ενιαίας αγοράς και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες πολιτικές. Θεωρώ ότι αν πραγματικά θέλουμε μια πιο ενοποιημένη και ισχυρή ενιαία αγορά, αυτό θα πρέπει να επηρεάσει όλες τις πολιτικές που απαρτίζουν την ενιαία αγορά. Και αυτό ισχύει και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, δεν χωρά αμφιβολία. Μια τελευταία ερώτηση. Όχι, ευχαριστούμε πολύ.